δικαιοσύνη για την περίοδο 2014-2020. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Γκιόνς. Πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια, περίοδος 2014-2020, άρχεται ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Βίνκλερ. Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η έκθεση Βίγκλερ. Έκθεση Φράγα. Πρωτόκολλο Συμφωνίας Αλληλευτική Σύμπραξης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση. Σύσταση Steinruck. Σύμβαση της ΔΟΕ για την ασφάλεια κατά τη χρησιμοποίηση χημικών προϊόντων στην εργασία. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Σύσταση Ματιέ Ουγιόν. Καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων. Ψηφί υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, φωνές από κάτω. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Σύσταση Σόλτς για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται σύσταση Μορέιρα. Εισαγωγή βοήου κρέατος. Ψηφίπε. Κατά. Επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Δεν σηκώνεται χέρια. Λοιπόν, σύσταση Μορέιρα, επαναλαμβάνω, για τις εισαγωγές βοήου κρέατος. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύσταση Κοτινή. Πρωτόκολλο Συμφωνίας Αλληλευτικής σύμπραξη με την ακτή Ελεφαντοστού. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση ΜΑΤΟ. Εισαγωγέ ορισμένων προϊόντων αλίας της καναρίου νήσους. Ονομαστική είναι η ψηφοφορία και αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση να ράχω. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική εκκλήση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νέισκι. Το ίδιο θέμα για το Ταμείο πακοσμιοποίηση. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Κοσλόφσκι. Το ίδιο θέμα πάντα. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Έκθεση Γέγλε. Διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία με τον Καναδά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Swinburne πλαίσιο ανάκαμψη και εξυγίανση για τα μη πιστωτικά ιδρύματα. Ψήφι Κατά αποχέ εγκρίνεται. Έκθεση Νίβλερ. Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψήφι Κατά απόχέ εγκρίνεται. Έκθεση Δελκαστήγιο. Υπολογιστικό νέφος. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται έκθεση σε εδώ. Έκθεση εξολόγησης του Μπερέκ. ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Ρόντουστ, κοινή ελευτική πολιτική. Η τροπολογία παριθμών 1, τμήμα πρώτο γιατί είναι κατά τμήματα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου, με προκειμένο. Έκθεση Στίβενσον. Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Χωρίς τροπολογία. Εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου λοιπόν. Έκθεση Αρσένη. Βορειοατολικός Ατλαντικός. Από θέματα βαθέων υδάτων και αλίας σε διεθνή ύδατα. Λοιπόν, 131 τροπολογίες έχουμε της αρμόδιας επιτροπής. Θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 29 ε, τροπολογία κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 62, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 131. Ψήφιπε. Κατά αποχές, έλεγχος. Παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν κρίνεται. Και καταπίπτει η επόμενη. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της Επιτροπής. Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το σχέδιο. Ορίστε. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο, παρακαλώ, κύριο Αρσένη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει του άρθρου 57 εδάφιο 2 του κανονισμού θα ήθελα η τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα να αναβληθεί και να δοθεί η εντολή στην Επιτροπή μας να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτό που πρότεινε ο κύριος Αρσένης. Ψηφίπε. Α, ορίστε κυρία Φράγα παρακαλώ. Πείτε μου. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας ζητώ να ψηφιστεί τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Το Κοινοβούλιο, οι περισσότερες πολιτικές ομάδες έχουν υπογράψει ένα συμβιβασμό που βλέπετε ότι υποστηρίζεται από την πλειοψηφία. Δεν υπάρχει λόγος αναβολής τελικής ψηφοφορίας. Εχθές μποϊκόταρε το συμβιβασμό εισηγητή, σήμερα έχασε στην Επιτροπή Αλίας είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας ο συμβασμός και προτείνω να προχωρήσουμε στην ψήφιση του νομοθετικού ψηφίσματος. Ο Πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει κυρία Φράγα, σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτό που μας πρότεινε ο κύριος Αρσένης πρέπει να ψηφιστεί. Αν θέλετε, αν θέλει το σώμα να ακολουθήσει εσάς θα καταψηφίσει. Αλλά πρέπει να θέσω σε ψηφοφορία αυτό που ζήτησε ο κύριος Αρσένης, έτσι κι αλλιώς. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση του εισηγητού, του κυρίου Αρσένη, υπό την εξή έννοια. Ζητεί αναβολή της τελικής ψηφοφορίας. Ψήφι υπέρ της ε, προτάσεως του κυρίου Αρσένη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η πρόταση του κυρίου Αρσένη. Τσεκ φωνές από κάτω. Εντάξει, εντάξει, θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. I think Πέρας. Απερίφθη η πρόταση του κυρίου Αρσένη. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε συνεπώς το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Σε Πέρας. Εγκρίνεται η πρόταση. Σαμος, al Περνάμε τώρα στην έκθεση Γκαρντίνη για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ψηφίζουμε το μπλοκ 1 των τροπολογιών υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ε, καταπίπτει το δεύτερο μπλοκ, ψηφίζουμε το σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί. Διακόπτει ο πρόεδρος. Ναι, την πρόταση επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προτείνουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που έχει δύο τροπολογίες, 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε την τροπολογία 108 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Σε Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψήφια. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Σάντζες Πρεζέδο. Συμβάσεις πίστος για ακίνητα κατοικίας. Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Και την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Murphy για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές. Το πρώτο μπλοκ τροπολογιών 1 έως 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Και ψηφίζουμε την τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 13 αρχίζει η ψηφοφορία. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπάρχει μόνο 13. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το ψήφισμα, το νομοθετικό ψήφισμα. Ναι, έχετε το λόγο. Ο κύριος Μέρφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε με βάση το άρθρο 57 παράγραφος 2 θα ήθελα να μην ψηφίσουμε για, τον, για την νομοθετική έκθεση, ψήφισμα μάλλον, και να γίνει αναπομπή στην Επιτροπή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ο πρώτος τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να γίνει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Θα ψηφίσουμε την πρόταση του κυρίου Μέρφη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα, περνάμε στην επόμενη έκθεση, που είναι η έκθεση Γκρότε για τον χρόνο διεξαγωγής πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής. Ψηφίζουμε απευθείας την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, σύμφωνα με το αίτημα της κυρίας Χάση, θα ψηφίσουμε την πρόταση ψηφίσματος για την ανάκτηση του χαρτιού. Σύμφωνοι. Ψηφίζουμε καταρχήν την τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος για τα κριτήρια για να ορίσουμε πότε το ανακτηθέν χαρτί ε, δεν ε, αποτελεί απόρριμα. Κυρία Μαγκίνες. Η κυρία Μαγκίνες ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας βοηθήσω γιατί πρόκειται για την τελευταία σελίδα του κατάλογου ψηφοφοριών. Δεν ξέρω αν είναι απόλυτα σαφές. Είναι η τελευταία σελίδα. Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια, ε, κυρία Μαγκίνες, στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Ξέρετε τι ψηφίζουμε. Ωραία, θαυμάσια. Γνωρίζετε όλοι τι ψηφίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ε, ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Με πολύ μικρή διαφορά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ωραία. Ας ελέγξουμε την 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε. Ψηφίζουμε την πέντε υπέρ κατά, αποχές. Ωραία, σε ελέγξουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Οκτώ. Αρχίζει η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος, αλλά διορθώνει. Ψηφίζουμε. 8. Υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. 7. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 7. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτώ. Οκτώ τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι αρχίζει η ψηφοφορία για την οκτώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 9. Πέρας. Εγκρίνεται αυτή τη φορά. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της. Περνάμε στην ονομαστική κλίση απευθείας, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία, θα διακόψουμε τώρα. Ε, ο κύριος Αλαφράνκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να διακόψω, ήθελα απλώς να πω ότι δεν ε, ε, λειτουργήσε το μηχάνημά μου όταν ψηφίσαμε την έκθεση Φράγα και υπερψήφισα. Ωραία, αποκαταστάθηκαν τα πράγματα. Τώρα θα διακόψουμε την ψηφοφορία για την ε, πανηγυρική συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μαλή και στις 12.30 θα συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, ε, κύριε Πρόεδρε και ΤΑ είναι μεγάλη τιμή για μας ε, το ότι ε, μας δίνεται η δυνατότητα να σας καλωσορίσουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χώρα σας, το Μάλι, είναι μια χώρα πολύ σημαντική για μας τα τραγικά γεγονότα, τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Τα παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγης.